Ε, την εντολή από τις 18 Φεβρουαρίου του 2015 για το νέο μέλος επιτροπής αυτής. Δεν υπάρχει αντίρρηση, άρα εγκρίνεται εντολή